Σας ευχαριστώ. Σύμφωνα λοιπόν τα πρακτικά της 18ης, της συνεδριάσεως της 18ης, παρακαλώ, τι θέλετε κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Θα ήθελα να σας εφιστήσω την προσοχή σε ένα θέμα να εκπέμψουμε τη συμπάθειά μας του, στην αδελφότητα αλλιέων της Ιρλανδίας, οι οποίοι έχασαν πέντε συναδέλφους τους αλλιείς την περασμένη εβδομάδα στα ανοιχτά του Κόρκ. Ευτυχώς υπήρξε ένας επιζών, δυστυχώς όμως πέντε αποβίωσαν. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συσχετίσουμε το γεγονός αυτό και να ε, αποτίσουμε φόρο τιμής και σε αυτούς τους αλλιείς. Ευχαριστώ. Βεβαίω, συνάδελφε, συμφωνούμε απολύτω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε τη θλίψη μα και για την προκείμενη περίπτωση. Πρακτικά, λοιπόν. Κύριε Σίμψον, θέλετε να πείτε κάτι.